Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα αρχίσει η κανονική μας συνεδρίαση, γιατί μας πιέζει κάπως ο χρόνος. Monsieur Moncade, il n'entend rien. S'il vous plaît. Merci de bien vouloir prendre. Παρακαλώ καθίστε. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη συνεδρίασή μας τον κύριο Ρολάντας Κριστιούνας, τον ε, Υφυπουργό της Λιθουανίας για τις εξωτερικές υποθέσεις, αρμόδιο και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας ε, σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο κύριος Κριστιούνας θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει στις 11 γιατί έχει πτήσει. Οπότε θα πρέπει να τηρήσουμε πιστά το χρόνο. Τον ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώνει και θέλουμε αγαστή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Λιθουανικής Προεδρίας στα πλαίσια και του νομοθετικού και διοργανικού πλαισίου που ισχύει με την συνθήκη της Λισαβόνας στα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουμε πολλές και συγκεκριμένες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν τις διαπραγματεύσεις για το Σώμα των Ευρωπαίων Εθελοντών για την ανθρωπιστική βοήθεια που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον και ανυπομονησία τις προτεραιότητες της Λιθωνικής Προεδρίας στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, Επίση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ανταλλαγή απόψεων θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο σε θέματα ανθρωπιστική βοήθειας ε, στο πλαίσιο της εκπεριτροπής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευρύτερα θέματα αναπτυξιακά και άλλα θα εξεταστούν στην ετήσια μας ε, συνεδρίαση με την Καθρίν Άστον, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τι εξωτερικέ υποθέσει και την πολιτική ασφάλεια και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, μα τίμησε με την παρουσία τη ε, τον περασμένο Μάιο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 20 λεπτά. E, parlamento Ναρέι, Man Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για εμένα σήμερα να σας παρουσιάζω τις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας μας στο θέμα της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κυλήσουν τα πράγματα Σωστά, τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά, εάν μου επιτρέπετε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στόχος της ανθρωπιστικής μας βοήθειας είναι η βοήθεια, η ανακούφιση, η προστασία για τα θύματα φυσικών ή ανθρώπινων καταστροφών σε τρίτες χώρες. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν πως πρέπει η ανθρωπιστική μας δράση να βασίζεται σε ανάγκες, να συμμορφώνεται με τις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Είμαστε υπερήφανοι για το ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός δόρητης και βασικός διεθνής φορέας ε, στο θέμα αυτό. Συνολικά η Ένωση και τα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύουν το 45% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για ανθρωπιστική βοήθεια παρά την ε, οικονομική κρίση η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αυξάνεται σταθερά. Σε μία πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ε, είχαμε σαφείς ενδείξεις πως ε, το 2011 η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν κάτι το οποίο υποστήριζαν 79% των Ευρωπαίων πολιτών και μέχρι το 2012 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί στο 88%. Βεβαίως ε, πρέπει πάντα να σκοπεύουμε να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε η βοήθειά μας να δίνεται με τρόπο στοχευμένο, με αρχές και βεβαίω να δίνουμε πάντα λόγο και στους πολίτες μας και στους ευπαθείς πληθυσμούς που θέλουμε να βοηθήσουμε. Έχοντας αυτά κατά νου χαράσουμε την πορεία του επόμενου εξαμήνου Προεδρία. Πριν κάνω την εισαγωγή μας λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ την προηγούμενη Προεδρία της Ιρλανδίας για τα επιτεύγματα της. Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη η οποία εφάρμοσε το πρόγραμμα του τρίου σε συνεργασία λοιπόν με την Ιρλανδία και με την Ελλάδα θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το ίδιο πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε σε τρεις ε, προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, με το Κοινοβούλιο για τον κανονισμό για ένα Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Δεύτερον, θα ξεκινήσουν συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ανθρωπιστικής βοήθειας και τρίτον σκοπεύουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ε, αντοχής ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ας ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν με το θέμα του θελοντισμού. Θεωρούμε πως είναι η πιο σημαντική μας νομοθετική πρόταση και βεβαίως ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ήδη υπάρχει κάποιος κοινός τόπος μεταξύ των θέσεων μας και σας βεβαιώ πως το Συμβούλιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η πρότασή μας να είναι υποφελής και για τους δικαιούχους και αποτελεσματική και να βασίζεται ε, σε πραγματικές ανάγκες και πραγματικά θεωρώ πως έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εσάς κυρία Πρόεδρε. Έχοντας κατά λοιπόν τις ευθύνες μας αυτές, η δεύτερη μας προτεραιότητα είναι να προχωρήσουν οι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής δράσης. Πρώτα απ' όλα αποτελεσματικότητα σημαίνει συντονισμός και βεβαίω πληροφόρηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπόν φορέων και μια συντονισμένη αντίδραση. Το βασικό μας έγγραφο πέρα είναι η συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το 2008 υιοθετήθηκε ένα πενταετές σχέδιο που συμπεριλάμβανε πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της συνένεσης αυτής. Θα υπάρξει μια αξιολόγηση και η τελική έκθεση αναμένεται τον Ιανουάριο του 2014. Βασικός στόχος είναι να υπάρξει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής και για να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση ανά τον κόσμο. Έτσι σκοπεύουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις μας και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται, οι προπολογισμοί μειώνονται, η παραβίαση του ανθρωπιστικού χώρου ε, δυστυχώς ε, επιδεινώνεται. Άρα πρέπει να συνεχίσουν οι συζητήσεις επί των ζητημάτων αυτών. Συνεχίζουμε λοιπόν να διασπείρουμε τις αξίες αυτές ε, της συνένεσης εντός και εκτός της Ένωσης. Ζητάμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια που είναι σαφώς υπέρ της ανθρωπιστικής δράσης με βάση κάποιες αρχές ε, να ε, μας βοηθήσει στη συζήτηση για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας. Και εδώ πέρα έρχομαι στην τρίτη μας προτεραιότητα που αφορά την αντοχή της πολιτικής μας αυτής. Όπως αναγνωρίζεται παγκοσμίω, η χρόνια φύση της φτώχειας ε, και η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών απαιτεί συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Τον Μάιο υιοθετήσαμε τα σχετικά συμπεράσματα στο Συμβούλιο και είπαμε πως η αντοχή αυτής της πολιτικής μας δίνει την δυνατότητα να υπάρξει ένας πολιτικός διάλογος και για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στη φάση εφαρμογής του σχεδίου η Προεδρία θα διευκολύνει τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το σχέδιό μας και τα μαθήματα που έχουμε αντλήσει από τις πρωτοβουλίες ΣΕΡ και ΑΖΙΡ. Επίσης, θα υπάρξει ένα φόρουμ ανταλλαγών απόψεων. Θα εξετάσουμε την κατάσταση σε διάφορες χώρες. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στο θέμα του συντονισμού. Ζητάμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει και αναμένουμε τον διάλογο επί του θέματος στους επόμενους 6 μήνες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάποιε τρέχουσε κρίσεις. Το πρώτο που σκέφτεται κανεί βεβαίω είναι η Συρία. Δύο έτη εμφυλίου πολέμου σημαίνουν πω υπάρχει μια ανθρωπιστική καταστροφή. Με τη βία βεβαίω ε, και αυτά τα οποία υφίστανται τα εκατομμύρια αμάχων. Οι άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες ε, είναι τεράστιες. Ο, ο ΙΕ θεωρεί πως χρειάζεται 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια είπα ε, Ένα δισεκατομμύριο από αυτά δεν έχει διατεθεί. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 678 εκατομμύρια ευρώ, όπως ξέρετε, και έχουμε δεσμευτεί για άλλα 400 εκατομμύρια. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ε, μια, οργανισμός με έναν ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της και στα δύο μέτωπα και στην προσπάθεια για να βρεθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση. Ζητάμε λοιπόν από όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις ανθρωπιστικές αρχές, το ανθρωπιστικό δίκαιο και να διευκολύνουν την παροχή βοήθειας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασχολείται κατά προτεραιότητα με τη Συρία. Όμως, ενώ δικαίως δίνεται προσοχή στη Συρία, δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλες περιοχές του κόσμου, όπως ο κόσμος υποφέρει και πεθαίνει λόγω συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών. Η Προεδρία μας βεβαίω θα ε, διεξαγάγει συνομιλίες ε, και για την κατάσταση σε χώρες όπως το Μαλί, την ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, Δημοκρατική, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Αιτή, αλλά και κάποιες ξεχασμένες κρίσεις όπως το Πακιστάν, τη Μιανμάρ, Βερμανία κτλ. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να επαναλάβω τη διάθεσή μας για στενή συνεργασία με την Επιτροπή σα Με βάση τις αρχέ που ανέφερα, όπω βλέπετε, είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για του επόμενου έξι μήνε. αλλά γνωρίζουμε πω έξι μήνε είναι απλά ένα βήμα στην πορεία μα. Και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει και σα ευχαριστώ για την προσοχή Σα euh, Σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές, τα μέλη της ομάδας ε, και δράτω με τις για να λάβω πρώτη εγώ το λόγο. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Χαίρομαι για την μελλοντική μας συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το Σώμα Ευρωπαίων Εθελοντών για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Θα αρχίσουμε το τριμερή διάλογο αρχές Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι ομόφωνα εγκριθήκε η έκθεσή μου για τη διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιση των διαπραγματεύσεων. Εμείς θα θέλαμε αυτό το σώμα να είναι αμυγός ε, ανθρωπιστικό, με πραγματική και γνήσια προστιθέμενη αξία. Ακόμη όμως δεν γνωρίζω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τη θέση του Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά την πρικοδότηση αυτού του σώματος Ευρωπαίων Εθελοντών για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις τραγικές ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου. Ε, η Συρία είναι η πιο εμφανής περίπτωση. Ήμουνα στο Μαλί πρόσφατα, θα επιστρέψω στις 28 Ιουλίου για τις εκλογές. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο βόρειο Μαλί είναι εξαιρετικά ανησυχητική και σοβαρή και έχει επισκιαστεί από την προεκλογική διαδικασία. Καλό θα ήταν λοιπόν να οργανωθεί μια ανταλλαγή απόψεων για το Μαλί προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Εσείς τι γνώμη έχετε για την πρόταση. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Πρώτα, ο λόγος στον κύριο Ντόνσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα αγγλικά και μετά λιθουανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε Υπουργέ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Θα ήθελα να κάνω πρώτα κάποιες παρατηρήσεις στα αγγλικά και να ολοκληρώσω μετά στα λιθουανικά. Καταρχήν εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για την έναρξη της Λιθουανικής Προεδρίας. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα και πολυάριθμες προκλήσεις και για την ανθρωπιστική βοήθεια και ως προς άλλα τμήματα του αναπτυξιακού πακέτου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο πτυχές. Είδαμε τι έγινε με την κρίση του ευρώ. Επιδεινώθηκε η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι μεγάλη πρόκληση για μας όχι μόνο να συνεχίσουμε το ρόλο μας ως δωρητού, αλλά να επιμείνουμε στη δέσμευσή μας ε, υπέρ της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Γιατί βλέπουμε ότι όπου επιδεινώνεται η οικονομική κατάσταση, έχουμε άμεσες και αρνητικές συνέπειες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι η Λιθουανία θα επιτύχει σε αυτό να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες και οι ιστορικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Η Λιθουανία δεν είναι ένας πολιτικός παράγοντας που θα έχει σημαντικό ρόλο για την υποσαχάριο Αφρική. Αλλά για άλλες περιοχές του κόσμου, την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, εκεί η Λιθουανία θα είναι πραγματικά σημαντικός ε, φορέας ε, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης. Η συνεργασία θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Θα πρέπει όμω πάθηση στη θυσία να αποφύγουμε τη δημιουργία πολιτικού κενού σε χώρε όπου η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται ακριβώ εξαιτία ε, τη διακοπή ή τη αναποτελεσματικότητα των ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Καλωσορίζω ε, εγκάρδια τη Λιθουανική Προεδρία και πιστεύω ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι κατεξοχήν ο τομέα που θα έχει πολλά να πει και να μάθει ε, και προ το δικό τη συμφέρον αλλά και προς όφελο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος λίγα λόγια και στα λιθουανικά. Ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά γιατί βρισκόμαστε εδώ στην αρχή της Λιθουανικής Προεδρίας, στην Παρθενική Προεδρία για τη Λιθουανία και με ιδιαίτερη συγκίνηση εύχομαι καλή επιτυχία στην πατρίδα μου. Στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε αυτό το πρόγραμμα με τις δυνατότητες που έχει η Λιθουανία να αποτρέψει τη δημιουργία πολιτικού κενού σε περιοχές του κόσμου που δεν είμαστε αρκετά παρόντες ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν εκεί πολιτικά κενά που θα καλυφθούν από μη δημοκρατικές δυνάμεις. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Λιθουανία για την Προεδρία της. Ο κύριος Λάστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως ε, για τη δυνατότητα αυτή για ανταλλαγή απόψε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη Λιθουανία που θα φιλοξενήσει σε λίγες μέρες την Λατιναμερικανική συνέλευση Ευρωλάτ και θεωρώ ότι η Λιθουανία ενδιαφέρεται να γνωρίσει από κοντά την ε, Λατινική Αμερική και το μήνυμα αυτής της διοργάνωσης είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σημεία που είναι και σημασία κατά τη γνώμη μου, όπως το σώμα των Ευρωπαίων Εθελοντών. Το επισημάνονται ως προτεραιότητα της Λιθουανικής Προεδρίας άλλωστε. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι ένα από τα θέματα που μπορούν να προωθηθούν στη διάρκεια της Λιθανικής Προεδρίας και να διεκπαιρεωθούν. Και χαίρομαι που το τονίσατε στην παρέμβασή σας. Το θέμα της αντοχής είναι σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο και στο θέμα αυτό της αντοχής. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που αποτελεί προτεραιότητα και για σας. Σε ό,τι αφορά τις, ανα, τους αναπτυξιακούς στόχους της Δύο σημεία είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά. Καταρχήν, οι προτάσεις μας μέχρι το 2015 και οι δράσεις μας μέχρι το 2015. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας ώστε να έχουμε το 2015 τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με το 2015 και μετά. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του βασικού μας στόχου που είναι η εκρίζωση της φτώχειας. Άλλωστε θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη για το θέμα αυτό το Σεπτέμβριο. Επίσης ε, το θέμα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η πρόοδος στο μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας θα έχει κεφαλαιώδη σημασία και εκεί ο ρόλος της Λιθουανικής Προεδρίας θα είναι νευραλγικός. Θα ήθελα παρακαλώ να λάβετε υπόψη και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πολύ δημοκρατικές και εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να δείξετε ευαισθησία απέναντι στι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία που θα εκπροσωπεί το σύνολο των, Ευρω... των Ευρωπαίων πολιτών. Και να ολοκληρώσω μια έκκληση που απευθύνουμε συστηματικά σε όλε τι προεδρίε. Θα ήθελα η Προεδρία σα να βρεθεί κοντά στην κοινωνία των πολιτών και κοντά στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό στη διάρκεια τη Προεδρία σα να αναπτυχθεί το αίσθημα της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι η Λιθουανική Προεδρία είναι πραγματικά στο πλευρό τους. Γιατί και η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σημαντικοί φορείς και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία, αλλά και του πρωταρχικού στόχου που είναι κοινό για όλου μα και που είναι ε, η εξάλληψη τη φτώχεια. Σα ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και θα είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Um, Μισό λεπτό, συντονιστή τη μεγαλύτερη ομάδα, <clears throat> θα ήθελα να μου επιτραπεί να πάρω το λόγο. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Το 64% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει επηρεαστεί από το 22 από φυσικές καταστροφές. Ας αναφερθούμε στην ΑΕΤ. 1,3 εκατομμύρια άτομα πέθαναν. Αυτό το έγγραφο είναι μια αναφορά των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μείωση των καταστροφών, του κινδύνου καταστροφών. Εδώ λοιπόν έχουμε τους στόχους ε, σαφώς ε, περιγραμμένους ε, Σας λέω από το στην σας διάταξη. Είπαμε να πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Είπαμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Όχι μόνο εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και εξοικονόμηση ε, ζώων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδρούμε εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε να κάνουμε ε, με κάτι που θα μπορούσαμε να εντάξουμε άμεσα στα προγράμματά μας. Ένα άλλο θέμα που αφορά το, το θέμα του φύλου. Ένα σημαντικό θέμα γι' αυτό το, το Κοινοβούλιο. 200 εκατομμύρια γυναίκες είναι πλήττονται στον κόσμο γιατί υπάρχουν, γίνονται διακρίσεις. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το συμπεριλάβετε στην μερισία διάταξη. Τώρα σε ό,τι αφορά το συντονισμό των συντονιστών. Εγώ είμαι ο συντονιστής για τον συντονισμό των δωρητών. Η Επιτροπή υπολόγισε ότι θα μπορούσε να γίνει εξοικονόμηση 6 δισεκατομμυρίων το χρόνο αν υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως είναι δύσκολο να επιτύχουμε το στόχο μας, είναι μεγάλο το ποσό Έχουμε μία έκθεση εδώ που μας δείχνει πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε 800, ε, ε, ε, εκατομμύρια ευρώ σε μία περίοδο λιτότητας, γιατί δεν το κάνουμε. Τι κάνουμε για να το βάλουμε στην ημερησία διάταξη. Το Συμβούλιο Υπουργών λέει ότι και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβληματίζονται για το θέμα του συντονισμού των δωρητών. Φανταστείτε γιατί η εξοικονόμηση μιλάνε 30 δις. Ε, ε, κάντε μια σύγκριση με τον προϋπολογισμό. Για σκεφτείτε, θα μπορούσαν να σωθούν ανθρώπινες ζωές με αυτά τα χρήματα. Θερμή παράκληση λοιπόν. Πέστε μου, θα προσπαθήσετε να προωθήσετε κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας το θέμα αυτό του συντονισμού των δωρητών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for all. πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ σχετικές οι ερωτήσεις που κάνετε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω απαντώντας στην κυρία Πρόεδρο. Βεβαίως είναι προτεραιότητα για μας η ενίσχυση των θελετών ε, έχουμε μία διασύνδεση και με τον προπολογισμό αυτής της νέας πρωτοβουλίας. Όπως τόνισα στην παρουσίασή μου, θα γίνει μια κοινή συζήτηση και ελπίζουμε να μπορέσει να περατωθεί αυτή η συζήτηση. Διεξάγεται και μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό και διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει βήματα για να περιοριστεί η αρχική πρόταση που έγινε από την Επιτροπή. Δεν είναι εύκολη βεβαίω η επιλογή από πλευρά τη Επιτροπή και δεν είναι εύκολη η επιλογή για το Συμβούλιο. Ξέρετε βεβαίως και εξάλλου αρκετοί από εσά το ανέφεραν ήδη ότι διανύουμε εποχές λιτότητας και αυτές οι εποχές μας υποχρεώνουν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και για το τελευταίο ευρώ που δαμβανάτε και Διαπιστώνουμε με χαρά ότι υπάρχει τάση αύξησης 2,8% Είναι λοιπόν επίτευγμα αυτό. Αν κοιτάξει κανείς ε, τα βασικά στοιχεία του ε, προϋπολογισμού. Δεν είναι ε, μυστικό ότι πετεύθη μια πολιτική συμφωνία και είναι για 30 εκατομμυρία λιγότερο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ορισμένες περικοπές. Δεν μπορούμε να, έχουμε, να τα ίδια με λιγότερα χρήματα σε όλους τους τομείς. Χαίρομαι ο, ο προϋπολογισμός για την ανάπτυξη αργά αλλά σταθερά αυξάνεται. Βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε μερικές ε, περικοπές. Τόνισα εξάλλου ότι οι ανάγκες αυξάνονται. Υπάρχει μια πρόταση να μειωθεί ο προπολογισμό για τους ε, κατά 147 νομίζω ότι είναι σημαντική η μείωση από το αρχικό ποσό. Μιλάμε για μείωση γύρω στο 30-40%. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μία πρωτοβουλία προς έγκριση θα έλεγα ότι είναι μια εξισορροπημένη πρόταση και στο Συμβούλιο πραγματικά πιστεύουμε ότι η προσπάθεια διατήρησης του ανθρωπιστικού προϋπολογισμού είναι κάτι, είναι κάτι για τον προϋπολογισμό στο σύνολό της. Αυτή είναι η στάση που υιοθετούμε στο Συμβούλιο. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μάλι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις. Όλοι μας περιμένουμε τις ε, εκλογές. Βεβαίως συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το τι έγινε σε αυτή τη χώρα. Όταν ξέσπασε η κρίση στο Μάλι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στηρίζοντας τη χώρα. Υπάρχουν κονδύλια, υπήρξαν για το 2013 και για το 2014. Δεν θεωρούμε <clears throat> την υπόθεση λήξασα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες, να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη. Αν θα μπορούσα να συνεχίσω και να απαντήσω στον ε, συμπατριώτη μου, τον κύριο Ντόνσκι, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ. Έχετε δίκιο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η ανθρωπιστική βοήθεια από τη φύση της αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφορά την παροχή βοήθεια σε ανθρώπους έτσι ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα. Όταν μιλάμε για καλύτερο συντονισμό μεταξύ της ε, βοήθειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι συνδέονται άμεσα αυτά τα θέματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μία έκτακτη βοήθεια. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί όταν συνδυάζουμε αυτά τα δύο, να υπάρχει μία μακρόπνοη πολιτική. Όταν ε, υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε προοδεύουν και τα πράγματα σε επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. Έχετε λοιπόν κύριε Ντόνσκι την ε, απόλυτη στήριξή μου στις απόψεις σας. Πραγματικά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. να αναφορά στην Ποσαχάρια Αφρική και στο τι θα μπορούσε να κάνει η Λιθουανία. Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει κάτι. ότι όχι άμεσα. Δεν θα έχουμε ένα παρελθόν και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει ε, πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε και μία πρόσφατη εμπειρία εντυπωσιακών αλλαγών. Δηλαδή οικονομίες με μία ε, κλειστή οικονομία. Τώρα περνά σε μια ελεύθερη οικονομία. Αυτή η εμπειρία θα έλεγα είναι καινούρια και θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε πολλές αφρικανικές χώρες. Γιατί πιστεύω ότι είναι αδύνατο να μιλάμε για προσαρμοστικότητα ε, στην εξέλιξη ή δυνατότητες αλλαγής της κατάστασης. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω απαντώντας τον κύριο Κόρτες Λάστρεμ. Αναφερθήκατε σε μία σειρά από σημαντικά θέματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι όλα πολύ σημαντικά για την Προεδρία μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2015 πλησιάζει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρώτο πυλόν το 2015 να κάνουμε ορισμένα πράγματα πριν από την ημερομηνία αυτή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Να δούμε όμως γιατί θα γίνει μετά. Και τα δύο αυτά συστατικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η συζήτηση για το τι θα συμβεί μετά το 2015 θα πρέπει να εξισορροπήσει και τις δύο πλευρές. Τι κάναμε στο παρελθόν, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Μετά το 2015. Βεβαίως οι προτεραιότητές μας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αφορούν την προετοιμασία για τη συνάντηση της Νέας Υόρκης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε στοιχεία σχετικά με το πώς αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και βεβαίως θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε αν υπάρχει ανάγκη συντονισμού ως προς τα διάφορα θέματα. Η προσαρμοστικότητα, αυτό είναι ένα θέμα που θίξατε ήδη. Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. Η προσαρμοστικότητα όταν τα χρήματα δεν περισσεύουν αποτελεί ένα μέρος της απάντησης. Βεβαίως χρειαζόμαστε έναν καλύτερο συντονισμό. Αυτό Νομίζω ότι με μικρές επενδύσεις καταφέρουμε να ε, εξοικονομήσουμε πολλά. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε σε αυτό το μέτωπο. Σε ό,τι αφορά το ECI, Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ACI, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας, ε, ξέρω ότι η συζήτηση είναι πολύ δύσκολη μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας όταν συμμετέχουμε σε αυτές τις θεσμικές συζητήσεις έχουμε πάντοτε στο νου μας ε, την Ευρώπη. Όλοι δουλεύουμε για την Ευρώπη. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από το τέλος του χρόνου. Γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ κακό το μήνυμα που θα σταλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους εταίρους της, ότι δεν είμαστε ικανοί να συμφωνήσουμε επί ενός νομικού πλαισίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια και πραγματικά είμαι αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την ε, βαρύτητα, τη σημασία των ΜΚΟ, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Σημαντικό ο ρόλο του στην ε, κοινωνία μα. Αυτή είναι η βασική ιδέα, να δράσουμε εκ των προτέρων, να, υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπτηση και η ΜΚΟ είναι το μέσον για να γίνει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα σημαντικές λοιπόν. Ο κύριος Μίτσος. Το ερώτημα του κύριου Μίτσου. σε ό,τι αφορά την ε, μείωση του κινδύνου καταστροφών πολύ σημαντικό θέμα και εκεί χρειάζεται αντοχή και προσαρμοστικότητα. Πώς θα μπορούσε κανείς ε, να θίξει αυτό το θέμα χωρίς ε, να αναφερθεί στο θέμα της μείωσης των κινδύνων. Για μας ε, είναι προτεραιότητα το θέμα της αντοχής και βεβαίως το θέμα της μείωσης των καταστροφών. Σε ό,τι αφορά το θέμα του φύλου, Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο σε αυτό το μέτωπο, αλλά η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και τα δικαιώματα των δύο φύλων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κανένας βεβαίως δεν αφισβητεί ότι θα είναι ε, προτεραιότητα. Ε, ναι, συγγνώμη όμως, εγώ αναφέρομαι στην δολοφονία γυναικών, στην δολοφονία ανθρώπων λόγω του φίλου τους. Όπως σας είπα, μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι να υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων στα... μεταξύ μας. Βεβαίω, η, η, που βρίσκεται εδώ δίχως άλλο θα εκφράσει και κύριοι τι απόψει της σε γενικά τα θέματα που αφορούν το φύ, τα δύο φύλλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας. Ενδεχομένω ορισμένα θέματα ε, θα συζητηθούν εκτενέστερα. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων, σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι η προτεραιότητά μας είναι ο συντονισμός, είναι η καλή... καλύτερη και πιο ενιαία εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Νέιζερ και μετά στον κύριο Χρύσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτά τα οποία είπατε. Χαίρομαι για τον ρεαλισμό σας και για τον στόχο αυτό που έχετε για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Θεωρώ πως ε, μέχρι το τέλος του 2014 θα θέλαμε κάτι το συγκεκριμένο. Η εθελοντική αυτή υπηρεσία είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό για όλους νέους και γέρους. Παράκλησή μου είναι να εκμεταλλευτείτε την τεχνογνωσία πολλών ΜΚΟ που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. και να διευρύνεται ίσως την ε, εμπειρία. Δεύτερη ερώτηση αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά το 2015 και θεωρώ πως θα πρέπει νομίζω να συμπεριλάβουμε και την αηφορία στόχους αυτούς. Χτες συζητήσαμε σε ένα άλλο πλαίσιο την πρόσβαση στην ενέργεια στην υποσαχάρια Αφρική και νομίζω πως αυτό είναι σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Καλό θα ήταν να συμπεριλάβετε την ε, ανανεώσιμη ενέργεια στους στόχους αυτούς. Τρίτη παρατήρηση αφορά την οτροπία δωρητών των κρατών μας. Είχαμε υποσχευθεί στις αντισόμενες χώρες να δίνουμε 0,7% του ΑΕΠ μας για αναπτυξιακή βοήθεια. Τα περισσότερα κράτη-μέλη απέχουν πάρα πολύ. Αντί για 0,7% η Γερμανία έχει μία θέση στο μισό. Και η χώρα σας επίσης. Τι πρέπει να κάνουμε για να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη τη δέσμευσή τους για αυτό το 0,7%. Και τελευταία παρατήρηση. Εντάξει μπορεί να ακούγεται κάπως δασκαλίστικο, αλλά μιλήσατε για τρίτο κόσμο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη διατύπωση γιατί ε, θεωρητικά έχουμε μια συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιος είναι ο τρίτος κόσμος, δηλαδή υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Ε, έχουμε μια αναπτυξιακή συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κόσμος είναι ένας. Σα ευχαριστώ κύριο gracias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, Λιθωνό Υπουργό για την πρώτη Λιθανική Προεδρία και σε λίγες μέρες ε, θα πάω στο Βίλνιους στην ε, Ισομερή Συνέλευση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Λατινοαμερικανικών Κοινοβουλίων Eurolat και εκεί θα μιλήσουμε και για τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική δεν ξέρω αν δεν ήμουν αρκετά συγκεντρωμένος στην ομιλία σας, αλλά αν δεν κάνω λάθος παραλείψατε τη Λατινική Αμερική. Ενώ και η περιοχή αυτή έχει πολλές ανάγκες, χαρακτηρίζεται από πολλές ανισότητες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Ποια είναι η γνώμη σας κύριε Υπουργέ για το θέμα αυτό. Βέβαια είναι μακριά η Λατινική Αμερική από τη Λιθουανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραγωνιστεί τελείω από τι λιθουανικέ προτεραιότητε. Η Ισπανία, αλλά όχι μόνο, ανησυχούν ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα. Είναι, από... είναι μία από τι συγκρούσει που έχουν αποκτήσει πια χρόνιο χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να πέσουν στη λύθη τέτοιου είδου χρόνια συγκρούσει. Επίση, συνεργασία με την Κίνα. Η διείσδυση της Κίνας στην Αφρική αλλά και στη Λατινική Αμερική είναι χαρακτηριστική. Η Κίνα καταβάλει προσπάθειες και αρχίζει και επεκτείνεται και στο θέμα της ε, συνεργασίας και κάνει επενδύσεις στις περιοχές αυτές. Όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, η Ευρώπη είναι ο πρώτος δωρητής ε, αναπτυξιακής συνεργασίας στον κόσμο και μερικές φορές χάνουμε πολύτιμες επενδυτικές ευκαιρίες που είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις μας για τους ε, Ευρωπαίους εργαζόμενους. Τις θέσεις αυτές και τις ευκαιρίες αυτές κερδίζει η Κίνα, παρόλο που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρόλο που δεν απασχολεί στα επενδυτικά της προγράμματα τοπικό πληθυσμό. Ποια είναι η θέση της Λιθανικής Προεδρίας ε, για αυτό το πρόβλημα. Κύριε Κορτές Λάστρα, ούτε ένα λεπτό δεν έχετε, γιατί θα προλάβει να απαντήσει ο Υπουργός. Λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση της ομάδας μας για τα θέματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Εμείς διαφέρουμε στην προσέγγιση μας από το ΕΛΚ. Εμείς θεωρούμε ότι τα σεξουαλικά δικαιώματα και τα δικαιώματα στην αναπαραγωγική υγεία ανήκουν στο ευρύ, στην ευρύτερη ομάδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Δεν νομίζω ότι κανένας αναφέρθηκε ε, στα θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Είναι ένα πολιτικό παίγνιο που διαρκεί εδώ και νέα χρόνια. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν εδώ για πολιτικά ωφέλη και ξεκίνησε από μια μη κυβερνητική οργάνωση. Εγώ μίλησα για τη φιλοκτονία. 200 εκατομμύρια γυναίκες αγνοούνται εξαιτία ε, άμβλωσης ε, λόγω του φύλου του εμβρίου και έχουμε εμβριοκτονίες και αυλώσεις που γίνονται ακριβώς επειδή τα έμβρια είναι θηλυκού γένους. Πώς μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει αυτό παρά μόνο φιλοκτονία. Αυτό είναι το θέμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο υπουργό είναι εύκαιρος μόνο μέχρι τις 11. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσει γιατί έχει αεροπλάνο στις Ξέρω ότι είναι διαφορετικά αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα απλώ να διαχωρίσω τη θέση μας από τη θέση του ΕΛ και τα θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, που κατά τη γνώμη των σοσιαλιστών είναι ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. from Mr. Ξεκινώ από την απάντηση προς τον κύριο Νόιζερ για τη βοήθεια στους εθελοντές. Πολύ σημαντικό το θέμα. Και επίσης είναι θέμα πώς θα αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη τα παγκόσμια θέματα και ελπίζω να θεσπιστούν οι νομοθετικές διατάξεις στη διάρκεια της ε, Λιθουανικής Προεδρίας για να προωθηθεί ο εθελοντισμός και να τεθούν και κάποιες προδιαγραφές για να εξασφαλιστεί και η προστασία των εθελοντών μας. Οι ΜΚΟ βοηθούν και παρέχουν τέτοια εθελοντική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ΜΚΟ και δεν θα αγνοηθεί καθόλου. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και το θέμα των δεξιακών στόχων της χιλιετίας, φυσικά είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να τονιστεί. Το θέμα της βιωσιμότητας της ε, ανθρωπιστικής μας βοήθειας είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει ε, να κάνουμε κάτι που δεν έχει συνέχεια. Η συνέχεια μας ενδιαφέρει και αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Επίσης, έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε κάποιους να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, αλλά θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο. Και αυτό σημαίνει βιωσιμότητα. Επίσης, ό,τι αφορά την οτροπία. Σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Είπατε ότι η Λιθουανία φαίνεται δεν υλοποιεί τους προηγούμενους στόχους. Εγώ συμμετείχα στις συζητήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θεσπίστηκαν οι στόχοι αυτοί πριν από αρκετά χρόνια. Και τότε εμεί ήμασταν νέα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε δεν ήταν το 0,7 ο στόχος αλλά 0,3. Φυσικά δύο είναι οι όψεις στο, στο νόμισμα πάντα και ε, όντως δεν έχουμε φτάσει ακόμα το 0,3 για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή είναι μία πλευρά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ε, και την άλλη πλευρά, ότι πολλές χώρες στη διάρκεια της κρίσης ε, χρειάστηκε να κάνουν περικοπές. Η Λιθουανία έκανε μια δημοσιονομική εξηγήση και κατάφερε ε, το δημοσιονομικό της έλλειμμα να το περιορίσει από το 9% στο 2,5%. Και κάναμε πολλές περικοπές, αλλά σας Διαβεβαιώνω ότι δεν κάναμε καμία περικοπή στην ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν την αυξήσαμε βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν την περικόψαμε, αλλά την διατηρήσαμε στο προηγούμενο επίπεδο. Κάτι που δεν κατάφεραν να κάνουν πολλές χώρες που ταλανίζονταν από την κρίση. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας βέβαια. Αν θυμάμαι καλά, μόνο 6 από τις 20 χώρες ε, κατάφεραν να υλοποιήσουν το στόχο του 0,7 της αναπτυξιακής βοήθειας ε. Εμείς έχουμε κάποιο δρόμο, Ακόμα είμαστε στο 0,3. Επίσης, στη διάρκεια της κρίσης προσχωρήσαμε σε διεθνείς οργανισμούς ανάπτυξης. Δηλαδή, συμβάλλουμε και εμείς τις πολυμερείς προσπάθειες για την ανάπτυξη στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τις χώρες του τρίτου κόσμου, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η διάκριση. Γιατί όταν εγώ λέω τρίτο, τρίτος. Ενώ τρίτες χώρες, όχι τρίτος κόσμος. Τρίτες χώρες, όχι χώρες του τρίτου κόσμου. Μπορεί εγώ να μπερδεύτηκα, αλλά όταν, εννοούσα, όταν έλεγα τρίτες χώρες, εννοούσα τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία περίπτωση τις χώρες του τρίτου κόσμου, υπανάπτυκτες, αναπτυσσόμενες χώρες. Κύριε Φίσας, Φυσικά με μεγάλη χαρά θα λάβω και εγώ μέρος ε, στην Eurolat γιατί θα καλυφθούν και εμπορικά ζητήματα. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε λοιπόν στο Βίλνιο, στα πλαίσια της Eurolat. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τη Λατινική Αμερική. Δεν αναφέρθηκα επί τούτου στη Λατινική Αμερική, αλλά σίγουρα έχουμε πολλές χώρες που εξαιτία της κρίσης κινδυνεύουν να μείνουν στη λύθη. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να θεωρήσει μεθοδολογίες για να μην ξεχαστούν κάποιες χώρες. Η Κολομβία, ας πούμε, είναι η προτεραιότητα στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ε, αναφέρθηκα λοιπόν ρητά στη Λατινική Αμερική από φόβο ξεχάσω κάποια συγκεκριμένη χώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για την περιοχή αυτή. Σίγουρα θα περιληφθεί στη συζήτηση και για το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία, για τα θέματα διαφοροποίηση και ούτω καθεξής. Εκεί σίγουρα θα αναφερθεί και η Λατινική Αμερική. Για την Κίνα τώρα Είμαι σε δύσκολη θέση εδώ, γιατί για πολιτικά θέματα αναπτυξιακής ε, συνεργασίας ε, αρμόδιο είναι περισσότερο η Λέιδη Άστον. Οπότε καλύτερα να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας προς την είπατε εκπρόσωπο που είναι αρμόδια για το πολιτικό σκέλος και φαντάζομαι στη συνεδρίαση που θα έχετε με την ε, είπατε εκπρόσωπο θα συζητήσετε και τα θέματα αυτά. Εγώ σας παρουσίασα τη θέση της Λιθουανικής Προεδρίας, ε, την εθνική περισσότερο θέση της Λιθουανίας, αλλά όχι τη θέση του Συμβουλίου. Αυτή θα σας την παρουσιάσει μάλλον η κυρία είπατε εκπρόσωπος, η κυρία Άσα. Για την σα, Δυτική Σαχάρα δεν είπατε τίποτα κύριε Υπουργέ. Για τη Σαχάρα έχετε, έχετε απάντηση για τη Δυτική Σαχάρα. Για να είμαι ειλικρινής, μου ξέφυγε μάλλον ε, η ερώτησή σας. Επειδή δεν θυμάμαι την ερώτηση, δεν θα ήθελα να απαντήσω. Αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση και ευχαρίστω να απαντήσω. Και ο κύριος ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Η Δυτική Σαχάρα, πρώην Ισπανική απικία, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Μαρόκου αυτή τη στιγμή. Έχει μετατραπεί σε χρόνια αυτό το πρόβλημα. Έχουμε στους καταβλισμούς του Τιντούφ στην Αλγερία χιλιάδες ανθρώπους. Βέβαια δεν βάζουν βόμβες γιατί δεν έχουν τρομοκρατική τάση και μερικές φορές τους ξεχνούμε ακριβώς επειδή δεν μετέρχονται βίας για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Αλλά είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση, καταπάτηση κατάφορη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνεργασία δυστυχώς ε, ε, έχει χαλαρώσει πολύ. Ακόμη και η Ισπανία που ασχολούνταν ιδιαίτερα έχει αποκοπεί από το θέμα αυτό. Άλλωστε η κατάσταση της Δυτική Σαχάρα συνδέεται άρρηκτα και με την κατάσταση του Σαχέλ. Πολύ φοβούμε ότι η Δυτική Σαχάρα είναι από τους μεγάλους λησμονημένους της πολιτικής μας. Γι' αυτό και σας απέφθηνα έκκληση κύριε Υπουργέ να μην ξεχάσετε την κατάσταση των Σαχαροϊτών και την δινή τους ε, ε, δινές συνθήκες διαβίωσης στους καταβλισμούς του Τιντούφ. Uh, λοιπόν, είναι διπλή η απάντηση. Όταν μιλάμε ε, για βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, οπωσδήποτε τίθεται το θέμα στο Συμβούλιο. Και έτσι πρέπει. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει πώς μας ενδιαφέρουν όλες οι κρίσεις. Γι' αυτό υπάρχει και ο όρος αυτός ξεχασμένη κρίση και έχουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και χαίρομαι που βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες ακριβώς περιοχές είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν ξεχνάει τίποτα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Αν μιλάμε επίσης και για πολιτικές αποφάσεις, και αυτά τα ζητήματα πρέπει να και τα ερωτήματα αυτά πρέπει να τα απευθύνετε στην ε, κυρία Άστον. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κατά το εξάμεινο της Λιθανικής Προεδρίας η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία μαζί σας για να βρούμε λύσεις ε, στα πολυάριθμα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και αναφέραμε και στη συζήτηση. Όπως είπε και ο κύριος Μιτσέλ πριν από λίγο, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είπατε και εσείς στην αρχή ότι είστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών, της διακρίσεις, τα προβλήματα των ηλικιωμένων και κάποια έκτροπα που γίνονται και παραβιάσεις σε αφρικανικές χώρες. Επίσης, διακρίσεις και σημαντική σημαντικές καταδίκες εις βάρος ομοφιλοφίλων και τα δικαιώματά τους θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και καλή επιτυχία στη Λιθουανική Προεδρία. Thank you. Merci, Alors, 11 heures. Qui Monsieur Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord, on va commencer. Alors nous allons euh, continuer, chers... collègues. Συνεχίζουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε καλέσει στην Επιτροπή μας τον κύριο Μαρκ Διμπούλ. Διμπούλ ή Διμπούλ εκτελεστικό διευθυντή του Παγκοσμίου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Θα εξετάσουμε τις ε, προτεραιότητες ε, του Παγκόσμιου Ταμείου για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές προτεραιότητε μετά τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει τη χρηματοδότηση του Ταμείου το Δεκέμβριο του 2011. Έκτοτε το Παγκόσμιο Ταμείο έχει εγκρίνει ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και θέτησε μια στρατηγική για την περίοδο 2012-2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη παρέχουν το 50% του συνόλου των πιστώσεων του Παγκοσμίου Ταμείου. Η Επιτροπή μας ε, δίνει μάχη για τις πολιτικές ε, της ανάπτυξης αλλά και της υγείας και από αυτήν την άποψη η καταπολέμηση του AIDS, της πηματίωσης και της ελονοσίας είναι σημαντικές μας προτεραιότητες. Το μέλλον θα είναι σημαντικό και τα επόμενα χρόνια για το Παγκόσμιο Ταμείο και θα πρέπει να ευθυγραμμίσει το πρόγραμμα εργασιών του με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους στόχους ηλιετίας και την ανάπτυξη για την περίοδο μετά το 2015. Έχετε κύριε Τιμπούλ το λόγο για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τις μεταρρυθμίσεις του Παγκόσμιου Ταμείου και το νέο μοντέλο χρηματοδότησης καθώς και τους μελλοντικούς στόχους της οργάνωσής σας. Έχετε το λόγο κύριε Ντιμπούλ, για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που μου δίνει χρόνο στην Επιτροπή σας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Παγκόσμιο Ταμείο και την στήριξη του Επιτρόπου του κυρίου Πίμπαλξ που φιλοξένησε την διάσκεψή μας και τον εκπροσωπούν σήμερα εδώ πέρα ο Κρίστιαν Σμιτ και ο Γιάν Πέιλερ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, δηλαδή ποιες είναι οι ευκαιρίες για το μέλλον για ε, HIV, φυματίωση και ελονοσία και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να πούμε κάτι που δεν είχαμε δει πριν από λίγα χρόνια. Έχουμε την πρόοδο της επιστήμης, της επιδημιολογίας και την τεράστια εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών για την εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων. Μπορούμε σήμερα να πούμε πως έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου των ασθενειών αυτών ως απειλή για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε μία μοναδική ευκαιρία. Και βεβαίως συναρπαστικό είναι πως με αυτά τα οποία μας λένε οι επιδημιολόγοι είναι πως πρέπει να αυτού αυτούς οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι και δεν έχουν δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί που κινδυνεύουν ιδιαίτερα ειδικά από φυματίωση και HIV είναι οι νεαρές γυναίκες, ε, ομοφιλόφιλοι άνδρες, ε, άνδρες ε, ε, και γυναίκες ναρκωμανείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα των ερωτικών υπηρεσιών. Οπότε είτε μιλάμε για Ευρώπη, Αφρική, Ευρασία και Κεντρική Αμερική, τα ζητήματα αυτά από πλευράς ε, ε, μπορούμε να τα δούμε μέσω του πρίσματος της ε, δημόσιας υγείας και να διευρύνουμε έτσι την τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι πως ε, δεν είναι λογικό να περιμένουμε χρόνια την ανάκαμψη των οικονομιών, γιατί βεβαίως οι μεταδοτικές ασθένειες δεν σέβονται τους προϋπολογισμούς και γνωρίζουμε από την Ουγγάντα πως μπορεί να επανέλθει ο HIV, βλέπουμε αύξηση των ποσοστών βλέπουμε πως εάν πιστοχωρήσουμε στην ελονοσία επανέρχεται αμέσως και στη φυματίωση πραγματικά υπάρχει ανισχυτική αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη, μέρη της Νοτιοαφρικής και ειδικά η φυματίωση που αντιστέκεται στα αντιβιωτικά ε, περνάει τα σύνορα. Και από το 2014 μέχρι το 2016 έχουμε μία ενίσχυση κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ελέγξουμε πλήρως αυτές τις ασθένειες τα επόμενα τρία χρόνια. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ρωτήστε συγκεκριμένα για το τι έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο. Με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε, όπως ξέρετε, έναν μετασχηματισμό που μας ε, επιτρέπει να έχουμε έναν προγραμματισμό για το μέλλον με μια εταιρική σχέση. Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο αναφέρατε, αντικατοπτρίζει τις ιδέες του 21ου αιώνα που δημιούργησαν το Ταμείο μας ε, με τη συνένεση του Μοντερέι, τη συμφωνία των Παρισίων, ε, τη συμφωνία του Άκρα και του Μπουσάν. Θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στις διάφορες χώρες και τους τομείς και τον ιδιωτικό τομέα. Προσπαθούμε δηλαδή όχι απλά να φτάσουμε μέχρι το τέλος των στόχων της αλλά και παραπέρα. Έχουμε εταίρους από τον ΟΗΕ, διμερεί προγράμματα, με τα κρατημέλη και την Κομισιόν της, ε, και την Κομισιόν την ίδια, κοινωνία των πολιτών, ε, οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, όλοι αυτοί για να προωθήσουμε την υγεία των ανθρώπων. Και όλα αυτά εντάσσονται σε μια εθνική στρατηγική υγείας, αντί να προωθούμε μια νέα στρατηγική υγείας. Και βεβαίως το άλλο θέμα είναι η προβλεψιμότητα, κάτι στο οποίο επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει, όπως είπα, προβλησιμότητα στη χρηματοδότηση. Και αντί για ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν στο δικό μας το πρόγραμμα και όχι στην εθνική στρατηγική των χωρών και οι χώρες δεν ήξεραν πόση ε, χρηματοδότηση θα είχαν, τώρα μπορούν να έχουν μια προβλέψιμη ροή πόρων για να μπορούν να προγραμματίσουν και να ξέρουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τους όρους αυτούς για να στηρίξουν τις εθνικές στρατηγικές υγείας. Το τρίτο στοιχείο είναι μια πλατφόρμα για να χρησιμοποιηθούν οι επενδύσεις για αυτές τις ασθένειες σε κάποια ευρύτερα συστήματα για να προωθηθεί όπως είπα η δημόσια υγεία. Εδώ υπάρχουν ευκαιρίες καθώς ε, τα ζητήματα αυτά αφορούν ε, πάρα πολλά άλλα ζητήματα όπως η αναπαραγωγική υγεία, η, η υγεία της μητέρας ε, και των παιδιών και των νεογέννητων και άλλες αρέστες. Και βεβαίως ε, για πρώτη φορά έχουμε αντιμετώπιση και πρόληψη των χρονίων ασθενειών σε κάποιες χώρες και άρα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για νέες ευκαιρίες όσον αφορά τη διαχείριση χρονίων ασθενειών επιπλέον επειδή κάποιες από τις επενδύσεις μας στον τομέα του HIV αφορά ειδικά τις γυναίκες νέες και ανήλικες υπάρχει μια πλατφόρμα για προγεννητική φροντίδα και αναπαραγωγική υγεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο συνολική προσέγγιση. Υπάρχει λοιπόν ένας νέος κύκλος χρηματοδότησης με βάση αυτές τις αρχές, την προβλεψιμότητα και την εταιρική σχέση με φοβερά αποτελέσματα. Ξέρω πως επισκεφτήκατε πρόσφατα τη Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουε ήταν από τις χώρες που ζήτησαν πρώτος χρηματοδότηση. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε ως εκστατική πραγματικά και την περιέγραψε ε, σαν να κάθονται δίπλα-δίπλα τα λιοντάρια με τους αμνούς. Υπήρχε δε και ο διάλογος που οδήγησε στις προτάσεις για την ε, Ζιμπάμπουε και Κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Μιανμάρ, μια χώρα η οποία όπως ξέρετε έχει κάποιες δυσκολίες ε, καθώς εκεί πέρα οι άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών με νέους τρόπους και, και εκεί πέρα εφαρμόσαμε τις αρχές που είπαμε, δηλαδή την επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε πως έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο με τις νέες αυτές προτάσεις έχουμε και ένα νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνου που δεν αφορά μόνο την ε, κατάχρηση των κονδυλίων όπου πλέον είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί και είχαμε τα νέα μέσα που συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση του Δουσού αλλά συζητήσαμε και το ζήτημα της κακής ή αναποτελεσματικής χρήσης των πόρων και αφιερώσαμε ανθρώπινους πόρους για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και για την επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, κοιτώντα πέρα από το 2015, με βάση τις αρχές που όρισε το πάνελ υψηλού επίπεδου που συμπεριλάμβανε και τον Επίτροπο Πίμπαλξ, έχουμε άρα κάποιες βιώσιμες προσεγγίσεις ε, για να δούμε τι θα γίνει με την υγεία, την επέκταση των δικαιωμάτων των γυναικών και τις ε, ευκαιρίες για τις νέες γυναίκες. Όπως ξέρουμε η εκπαίδευση και η υγεία είναι κάποια βασικά πράγματα που κρίνουν το εάν μια νέα γυναίκα θα είναι επιτυχής στην ε, κοινωνία και θα μπορέσει να έχει κάποιες ευκαιρίες. Εάν δούμε λοιπόν τις αρχές για την περίοδο μετά το 2015 καθώς έχουμε τη δυνατότητα να νικήσουμε αυτές τις ε, τρεις ασθένειες Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και αναμένουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της για να γίνει όλο αυτό πραγματικό. Του Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος ήθελε να πάρει το λόγο? <coughs> Monsieur Mitchell. Thank you, um, thank you, Chairperson. Um, um, in the area of sexual and reproductive health, um,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 I think if we had um, a graph here, we would see huge numbers for for, for women dying from heart attacks, women in particular, but women and men. Uh, τι ακριβώς κάνετε. Θα πρέπει να τύχουν τις ίδιες προσοχής και οι ασθένειες αυτές. Θα επιθυμούσαμε να γνωρίσουμε τι ακριβώς κάνετε. Μήπως θα μπορούσατε να ε, θέσετε και πάλι τις προτεραιότητές σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή έστειλε ένα, μία επιστολή την 4η Ιουλίου για να αφαιρθεί στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο Σιρλάνκα και στο Κολόμπου. Επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει την χρηματοδότηση πριν από δύο χρόνια. Από τότε την αναλάβαμε και πάλι λαμβάνοντας ε, στηριζόμενοι στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. Δίχως άλλο, υπάρχει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης που καθιστά τη χρηματοδότηση περισσότερο περισσότερο αποτελεσματική. Και αυτό αποτελεί απάντηση και στο ερώτημα του κυρίου Μίτσελ ό,τι αφορά το θέμα του συντονισμού για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Θα πρέπει δηλαδή το μοντέλο αυτό να ενσωματωθεί με έναν τρόπο που να επιτρέπει την παροχή όλων των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες, είτε μιλάμε για λοιμώδη είτε για μη λοιμώδη νοσήματα. Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μας δίνει τη δυνατότητα να μην περιοριζόμαστε μόνο σε αποφάσεις που λαμβάνονται στην Γενέβη να έχουμε άμεση συμμετοχή. Το Ταμείο παραμένει η Ταμεία για τις τρεις ασθένειες, αλλά βεβαίως έχει μια πιο ενεργό συμμετοχή όπου παίζουν κάποιο ρόλο όχι μόνο οι εντορητές στη Γενέβη και στις Βρυξέλλες, αλλά και οι ίδιες οι χώρες. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτό το σημείο Πιστεύουμε ότι αργότερα θα επανατροφοδοτηθεί το Ταμείο μέχρι το 2016 και η άποψη της Επιτροπής είναι ότι θα γίνει μία μελέτη τουλάχιστον ε, στα πλαίσια των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να, κρατήσουμε, να κρατηθούμε σε αυτό το επίπεδο για το άμεσο μέλλον. Δεν θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι η νέα ηγεσία του Ταμείου, του οποίου επικεφαλής ο κύριος Γκάιντερ, έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτού του χρονοδιαγράμματος. Κύριε Κορτές. Γνωρίζετε τη θέση μας για το έργο του Παγκοσμίου Ταμείου και ζήτησα το λόγο για να επαναλάβω και να ξέρω και πάλι το έργο του Παγκόσμιο Ταμείο, από τη γνώμη μας είναι αξιέπαινο και θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο αξιέπαινο και πολύ αποτελεσματικό. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί. Γνωρίζετε την υποστήριξη της ομάδας μας προς το Ταμείο, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η συμβολή σας στην αντιμετώπιση ασθενειών ε, είναι κέρια. Ο κύριος Νόιζερ. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Ταμείου. Ο κύριος Ντιμπούλ ε, ξεκαθάρισε νομίζω το ποιες ε, προοπτικές μας προσφέρει το Ταμείο αυτό και πόσο αποτελεσματικά εργάζεται για την καταπολέμηση των τριών αυτών ασθενειών και θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται εκεί. Είναι μοναδική η κατάσταση, δηλαδή ε, ιδιώτες ε, δωρητές ε, και δημόσιοι δωρητές έχουν χαράξει από κοινού μια στρατηγική αλλά βεβαίως για να συνεχιστεί αυτό χρειάζεται μια ασφάλεια στον προγραμματισμό η οποία υπάρχει τώρα με τις δεσμεύσεις μέχρι το 2016 αλλά χρειάζεται Χρειάζεται ακόμη περισσότερα λεφτά από τα κράτη-μέλη. Και εδώ πέρα υπάρχει η τάση κάποια κράτη-μέλη να παγώνουν τα λεφτά, να μειώνουν τα λεφτά. Το ερώτημά μου είναι με ποια στρατηγική ε, σκοπεύετε να αποκτήσετε περισσότερα κονδύλια η Γερμανία. Πόσο ξέρω πάγωσε τα ποσά που δίνει. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι ε, πολύ καλός δωρητής. Από την Ιταλία ακούμε πως ίσως αποσύρθει. Οπότε, ποια στρατηγική έχει το Παγκόσμιο Ταμείο για να επηρεάσει τα κράτη-μέλη. Και το άλλο ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένοι οι ιδιώτες, τα ιδιωτικά ιδρύματα να μπουν στο Παγκόσμιο Ταμείο αυτό και να διαθέσουν κονδύλια. Τέλος, στη συζήτηση με τις χώρες ΑΚΕ διαπιστώσαμε πόσο καλή είναι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Παγκόσμιο Ταμείο ε, και ποιες δυνατότητες υπάρχουν γιατί δεν είναι ίσως αρκετά ενημερωμένοι. Αναφέρθηκαν Επίσης ε, παραδείγματα αποτελεσματικής εργασίας, η Ζιμπάμπουε που το συζητήσαμε χθες, η Μιανμάρ. Θεωρώ πως ακριβώς το Παγκόσμιο Ταμείο έχει εδώ πέρα δυνατότητες που δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω θα πρέπει να διατηρηθούν αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Μάρκεντι Τιμπίλ για να ε, συμπληρώσει την παρέμβασή του. Ευχαριστώ πολύ για τα θαυμάσια αυτά ερωτήματα. Θα ήθελα να τα πάρω με τη σειρά. Σε ό,τι αφορά το μοντέλο των αδειών, αγοράζω, όλες μας οι αγορές αφορούν γενώσιμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο οι εταιρείε συμμετέχουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε θέματα που αφορούν την, ανθεκτη, την αντοχή. Πολύ λίγες χώρες έχουν νόμους ή ε, αντιοδότησης οι διεθνεί συμφωνίε ε, δεν αποτέλεσαν ιδιαίτερο πρόβλημα για μα. Σε ό,τι αφορά τα μη λοιμώδη νοσήματα, θα πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα. Το AIDS αποτελεί το βασικό αίτιο θανάτου για γυναίκε σε αναπαραγωγική ηλικία. Δεν αν δεν αντιμετωπίσουμε το AIDS δεν μπορούμε να έχουμε υγιείς γυναίκες. Η φυματίωση είναι μια ασθένεια που πλήττει τι εγγύου γυναίκε και τα μικρά παιδιά επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων εστιάζουν την προσοχή τους ε, εκεί γιατί ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στις χώρες τους αν πεθαίνουν οι νέοι άνθρωποι. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι ασθένειες αυτές που πλήττουν τους εργαζόμενους, τις μητέρες, τους πατεράδες τους δασκάλους, όλους ε, τους ανθρώπους τους οποίους βασίζεται η οικονομία και που αποτελούν θύματα AIDS και φυματίες. Όπως είπε ο κύριος Σμίτ, λόγω της, ε, του νέου μοντέλου προσέγγισης και χρηματοδότησης ε, και επειδή η πρώτη φορά που πραγματικά μας απασχολεί τόσο πολύ το θέμα έχουμε ένα μοντέλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αποτελεί αίτιο, θανάτου για πολλές γυναίκες στην Αφρική. Όπως είπε ο κύριος Σμίτ, δεν το χρηματοδοτήσουμε αυτό, αλλά υπάρχει μια βάση, μια υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρόνια παροχή ε, βοήθειας. Ο Κύριε Κόρτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Ευχαριστούμε για την στήριξη η δική σας και των συναδέλφων σας. Η στήριξή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Κύριε Νάσαρ, ευχαριστώ πολύ και εσάς για τα σχόλιά σας. Πιστεύω Και βεβαίως ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την υποστήριξη που μας παρέχετε. Η στρατηγική είναι το να θέτουμε τα θέματα όπως τα θέσαμε εδώ, αλλά υπάρχει μία ιστορική ευκαιρία ε, που αφορά την, τα ανθρώπινα δικαιώματα το θέμα είναι ότι αν ξεσπάσει κάποια επιδημία δεν έχουμε τα επισημονικά μέσα για να τις καταπολεμήσουμε. Χάνατε λοιπόν μία γενιά ολόκληρη. Όπως είπε ο φίλος μου, ε, τα σημερινά δεινά θα είναι και τα αυριανά δεινά. Ε, αναφέρεται αρκετές χώρες οι οποίες έχουν ε, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Ταμείο. Έχουμε και μία ε, νέα προσέγγιση. Δηλαδή δεν ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη αναζητώντας πόρους. Ε, έχουμε πολλούς πυλώνες που αφορούν πόρους και από άλλα μέρη του κόσμου. Έχουμε συμμετοχή και από την Αφρική το τομέα της καταπολέμησης του AIDS. Το ίδιο συμβαίνει και ε, σε ό,τι αφορά την φυματίωση και την ε, ελονοσία. Προς αυτή την, κυβέρνηση, την κατεύθυνση κινούμεθα. Προσπαθούμε να πείσουμε και τι κυβερνήσει να έχουν συμβολή. Μπορούν, δεν μπορούν να ζητάνε αύξηση των ε, πόρων όταν δεν συμβάλλουν και εκείνε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη όταν χάνουν ολόκληρε γενιέ από αυτές τις ασθένειες. Κινητοποιείται λοιπόν και η Αφρική και η G20 συνεργάζονται μαζί μας. Οι πόροι δεν θα είναι άμεση αλλά η συνεργασία μαζί τους και η συνεπένδυση θα βοηθήσει γιατί είναι χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία μας. Αναφερθήκατε στον ιδιωτικό τομέα μας, ε, απασχολεί ιδιαίτερα ο ιδιωτικός τομέας. Η Coca-Cola για παράδειγμα στην Ταζανία προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα σύστημα ε, ε, διανομής Έχουμε εταιρείε που συμβάλλουν άμεσα στο δικό μας ε, ε, ταμείο μέσω του product ε, web Ευελπιστούμε ότι θα, υπάρξουν, ε, θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ιδιωτικό τομέα. 65 εκατομμύρια, μας υποσχέθηκαν να, να δοθούν 65 εκατομμύρια δολάρια, 130 συνεπώς συνολικά εκατομμύρια δολάρια και με, κοιτάζουμε και αλλού. Δηλαδή <clears throat> προσπαθούμε και εμείς να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών μας. Βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος των πόρων θα χρειαστεί να προέλθει από τους παραδοσιακούς δωρητές. Και μέχρι τον επόμενο κύκλο θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια μεγαλύτερη αύξηση στις άμεσες εισφορές. Θέσατε πολύ σημαντικά θέματα και σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Σμίτ για τα σχόλια που έκανε. Ήταν εξαίρετη η συνεργασία με τον κύριο Σμιτ και τον κύριο Πέιλ ε, και ο Επίτροπος βεβαίως μας υποστήριξε. Θα ήθελα να τελειώσω ευχαριστώντας τον Επίτροπο, ευχαριστώντας για τις θαυμάσιε ερωτήσεις. Θα ήθελα να επίσης να πω ότι ένα πρώην μέλλον του Κοινοβουλίου, ο Σεράβισερ από τον Καναδά, βρίσκεται ανάμεσά μας. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε να πάρω μέρος σε αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για την ομιλία σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο Ταμείο κατά την εκτέλεση της αποστολής του. Αγαπητοί συνάδελφοι, μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας μετέβη στην Κολομβία 12 με 14 Απριλίου προκειμένου να εξετάσει δύο καθόδη ζητήματα, αυτό των εκτοπιστέντων και της απολωτρίας των γεών. Τέσσερις ευρωβουλευτές συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μας, ο κύριος Κόρτες Λάστρα, η κυρία Κατρίν Γκρέση, ο κύριος Δίας Δεμέρα και ο κύριος Σαντιάγκο Φίσας. Θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής αντιπροσωπείας, τον κύριο Κορτές Λάστρα, για να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της αντιπροσωπείας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε λίγοι βέβαια, λίγη και εκλεκτή, όπως λέμε, λέει η Πρόεδρος. Όντως, είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας Επιτροπής μας στην Κολομβία και ασχοληθήκαμε με τα θέματα που ενέκριναν οι συντονιστές, δηλαδή αξιολόγηση ε, και μελέτη το καθόδου ζητήματος των εκτοπιστέντων ε, προσώπων και της απαλωτρίωσης των γεών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για την ενεργό του συμμετοχή του, την Κατερίνη, τον Αγουστίν και τον Σαντιάγο, καθώς και την γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης, αλλά και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βογκοτά, γιατί μας παρήχε ανεκτήμητη βοήθεια σε ένα περίπλοκο και δύσκολο περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες οι Κολομβιανοί επλήγησαν τα μάλα από τις ένοπλες σειράξεις στη χώρα αυτή. Η επίσκεψή μας μάλιστα έλαβε χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ τη Κολοβιανή κυβέρνηση και των ΦΑΡΚ. Η ειρηνευτική αυτή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από μια συνεχή εσωτερική σύγκρουση, παρουσία ε, με συμμετοχή μάλλον των στρατιωτικών ε, δυνάμεων της Κολομβίας αλλά και παραστρατιωτικών και αντάρτικων δυνάμεων. Και μάλιστα η συνέχιση αυτή της ε, εσωτερικής ένοπλης σύραξης έχει τραγικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό, δηλαδή στους εσωτερικά εκτοπισμένους, στους πρόσφυγες, αλλά και στο σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Είχαμε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και υπερφορτωμένο. Είχαμε πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους ε, της κυβέρνησης, υπουργό, με τον Υπουργό Γεωργίας, ε, Δικαιοσύνης, ε, με τοπικές οργανώσεις, μέλη του, της Γερουσίας, των Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης είχαμε συναντήσεις με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και την ύπατη αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και μάλιστα στο Wagen Pass ε, παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καλή, στο Σανταντέρ, το Κιλατσάου. Είχαμε επαφές με τοπικούς γεωργούς, με κυβερνητικές οργανώσεις, με θύματα, οργανώσεις θυμάτων και τοπικές αρχές. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω τα βασικά συμπεράσματα της αποστολής μας. Καταρχήν, η Κολομβιανή κυβέρνηση εφαρμόζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπίσει και τις βαθύτερες αιτίε της ε, στρατηγική σύγκρουση, αλλά να καταπολεμήσει ταυτόχρονα την συνεχή ανεργία και την ε, μόνιμη φτώχεια, καθώς και την ε, επισφαλή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κατάσταση. Η κυβέρνηση Σάντος ε, ανέλαβε τη δέσμευση να ενισχύσει τον ρόλο της Κολομβίας στο διεθνές προσκήνιο και να συμβάλλει στην ε, διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων αλλά και τη βελτίωση των επενδυτικών σχέσεων. Συμφωνούμε λοιπόν με την παρατήρηση των διεθνών εταίρων ότι το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κολομβίας δημιούργησε ένα πρόσφορο κλίμα πολιτικό για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την ενευτική διαδικασία και να συνεχίσει την ανθρωπιστική τη βοήθεια. Κάτι που αναγνωρίστηκε από όλου του ενδιαφερόμενου. Και μάλιστα η έκθεση για την συνεργασία με την Κολομβία για το 2007-2013 αναφέρθηκε σε ποσό 160 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τονίσαμε την θετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συνέχιση της διμερούς σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας ε, καθώς και με, με τον Ισημερινό και το Περού. Χρειαζόμαστε μια συνεπή συνέχιση της βοήθειας και σταδιακή μείωση της ενίσχυσης προς τις χώρες μέσω εισοδήματο. Και μάλιστα το 2011 εγκρίθηκε από την κυβέρνηση ο νόμος 1448 που προβλέπει διάφορες μορφές αποζημίωσης καθώς και την οικονομική αποζημίωση και άλλα προνόμια όπως πρόσβαση στην παιδεία και στην υγεία. Αναφέρεται στο νόμο αυτό ποιες είναι οι διαδικασίες για, την επιστροφή των γεών στους εσωτερικά εκτοπισμένους και επίσης ε, την παράνομη κατοχή γεών από εγκληματικέ οργανώσεις. Η εφαρμογή του νόμου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και ε, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μια δεκαετία για να εφαρμοστεί πλήρως. Στις συνεδριάσεις μας ε, ακούσαμε πολλά σχόλια για τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου αυτού. Μερικοί συνομιλητές μας έκριναν ότι η παρουσία στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και η συνεχή σύραξη στις γεωργικές περιοχές εμποδίζει την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Επίσης υπάρχουν κενά στην επιμελητία αλλά και στην ασφάλεια και προστασία, ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες κάποιων συνηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την απογραφή των θυμάτων, την καταγραφή των καταγγελιών και των ατασταλιών και την διεκπαιρέωση κάποιων ερευνών για εγκλήματα. Πολλοί, πολλοί γεωργοί που, και χωρικοί που εκδιώχθηκαν από τα χωράφια τους διαμένουν αυτή τη στιγμή στις πόλεις και φοβούνται να επιστρέψουν στην Ήπεθρο γιατί λείπουν και οι υποδομές και επιπλέον φοβούνται την παρουσία παρακρατικών οργανώσεων. Άλλωστε η τρομοκρατία και το ραθρεμπόριο ναρκωτικών εξακολουθούν να απειλούν την ε, ασφάλεια και με βάση τις ε, εκτιμήσεις διεθνών και τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και το ΟΗΕ τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αντιμετωπίσουν στην Κολομβία σημαντικές προκλήσεις στο μέλλον. Οι κολομβιανές αρχές όμως θεωρούν ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που διευκολύνει την επιστροφή εγκαταλελειμμένων ή επεξερεμένων γεών και την διευκόλυνση επιστροφής των θυμάτων θα έχει κεφαλαιώδη σημασία. Ο νόμος αυτός 1448 αποτελεί ένα τμήμα ενός περίπλοκου πλαισίου μεταβατικής δικαιοσύνης που θεωρεί ότι σε περίπτωση ένοπλης σύραξης ε, και για την αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη φυσικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το ρυθμό εφαρμογής αυτού του νόμου, του 1448, ε, θεωρούμε ότι αυτό το νομικό πλαίσιο δίνει κάποια σημαντικά εργαλεία για την ανέβρεση μιας ε, ε συνεπούς λύσης για την επίλυση του κοινωνικο-οικονομικού προβλήματος της Κολομβίας. Τώρα, η στάση μας είναι η διατήρηση διμερούς συνεργασίας με Κολομβία, Περού και Εκουαδόρ και προσδιορισμό μιας ε, σταδιακής εξάλληψης ε, του, ε, της αναπτυξιακής συνεργασίας. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε την Κολομβία και να καταπολεμήσουμε την καλλιέργεια κοκαίνης, κόκας μάλλον, φύτου κόκας και να, πατάξουμε, βοηθήσουμε την Κολομβία να πατάξει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, να ενισχύσουμε το ρόλο της τοπικής οικονομίας, των ομάδων των γηγενών, των ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα σε περιοχές που επλήγησαν από την ένοπλη σύραξη. Να συνεχίσουμε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΕΚΟ, να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Διμερών Δωρητών και των Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Να βελτιώσουμε το διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να εξασφαλίσουμε να διαβεβαιωθούμε μάλλον ότι δεν θα χρηματοδοτούμε προγράμματα σε εγκαταλειμμένες γεές ή γεές που έχουν απαλωτριωθεί. Γιατί σε καμία περίπτωση θα πρέπει ε, να στηρίξουμε προγράμματα σε γεές που έχουν ε, υπεξαιρέσει ε, παραστατικές δυνάμεις. Επίσης θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα εργασιακών συνθηκών, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Η αντιπροσωπεία μας πραγματοποίησε πολύ σημαντική αποστολή και είχαμε και πολύ σημαντικό θεσμικό πρόγραμμα και ενημερωθήκαμε από πρώτο χέρι για το θεσμικό έργο της Κολομβίας αλλά είδαμε και η την πραγματικότητα στην Κολομβία την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάντως, στις συνεδριάσεις και συναντήσεις που είχαμε με πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με εκπροσώπους ε, των κρατών μελών αρμόδιους για θέματα συνεργασίας όλοι χωρίς καμία εξαίρεση τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης ε, της ε, συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κολομβία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κορτές Λάστρα. Εξαιρετική η παρουσίαση. Κύριε Φίσας, ζητήσατε το λόγο. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω σχεδόν τίποτα σε αυτά που μας είπε ο Ρικάρδο Κορτές Λάστρα. Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της αντιπροσωπείας στην Κολομβία και θα ήθελα να πω ότι από όλες τις αντιπροσωπείες και τις αποστολές που έκανα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή στην Κολομβία ήταν ε, η αποστολή στην οποία είχαμε τις περισσότερες συναντήσεις και την περισσότερη πυκνότητα επαφών στο πρόγραμμά μας. Δεν είχαμε σχεδόν ούτε λεπτό διακοπής και ανάπαυλας. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ε, τους αριθμούς, αλλά αναφέρονται περίπου 6 εκατομμύρια εκτοπισμένοι που εγκατέλειψαν τη, τα χωράφια τους, τη γη τους, εξαιτίας της βίας που επικράτησε, της ένοπλης σύραξης, των Αντάρτικων, των ΦΑΡΚ αυτή τη στιγμή εκτελήσονται διαπραγματεύσει μεταξύ της Κολομβιανής κυβέρνησης και των ΦΑΡΚ που γίνεται με θεματική διάρθρωση. Το θέμα της γεωργίας φαίνεται ότι διεκπαιρεώθηκε και επιλύθηκε το Μάιο. Βέβαια θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το πώς ε, η ειρηνευτική λύση θα επηρεάσει την ανακατανομή των γεών, γιατί ο νόμος είναι μεν καλός, αλλά είναι δυσεφάρμοστος, γιατί πολλές ε, οικογένειες χωρικών έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια τους ε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια και διαμένουν στις πόλεις και η επιστροφή τους είναι δύσκολη, ιδιαίτερα για τις οικογένειές τους, γιατί στερούνται στοιχειωδών υπηρεσιών, μου είδατος ε, εκπαίδευσης, υγείας. Η επιστροφή λοιπόν στις γέες τους, ακόμη και να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητάς τους, δεν θα είναι εύκολη. Γιατί το θέμα είναι να επιστρέψουν σε μια περιοχή που θα εξασφαλίσουν καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Και πολλά προβλήματα υπάρχουν ιδιαίτερα σε, στις ζώνες που έχουμε παράνομη εξόριξη ορυκτού πλούτου με πολυεθνικές που εκμεταλλεύονται παράνομα τον ορυκτό πλούτο της Κολομβίας και εφαρμόζουν συστήματα για την ε, ε, απαγόρευση της επιστροφής των γεών, ακόμη και όταν υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή και μας έκανε μια πολύ καλή σύνοψη των αποτελεσμάτων της ο πρόεδρος ε, Κορτές Λάστρα. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Νικόλ Μάρη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο βουλευτές για αυτά τα οποία μας είπαν σήμερα προφορικός που βεβαίως συμπληρώνουν και την γραπτή έκθεση που διαβάσαμε με ενδιαφέρον και καλωσορίζουμε τα ευρήματά σας και οι συστάσεις σας νομίζω πως ε, πηγαίνουν προς ε, το εκεί που προτείνουμε και εμείς. Ε, επίσης αξίζει να αναφερθεί πως πρέπει να εντατικοποιηθεί ο διάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πρώτη φορά είχε γίνει σε επίπεδο πρωτευουσών έγινε και στις ε, Βρυξέλλες ε, στις 17 Ιουνίου και με την ε, Κολομβία με όλες τις αρχές που είχαν πολιτικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες και με υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθαγενών φυλών και γνωρίζουμε βεβαίως την απειλή και από τις τον εξορυκτικό κλάδο και είναι γνωστό αυτό σε επίπεδο Λατινικής Αμερικής και προετοιμάζουμε κάποιες προτάσεις. Αλλά στην περίπτωση της Κολομβίας είναι σοβαρή η πρόκληση και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο πλαίσιο του προγράμματος ε, των του χωρών όλων και εξάλλου εμείς έχουμε τονίσει πως πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη πραγματική περίοδο. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει το λόγο όχι. Ωραία. Οπότε θα ξαναδώσω τον ε, λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και την ΕΕΔ και να πω δύο-τρία θέματα που κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ σημαντικά στο ταξίδι μας. Πρώτον, βρεθήκαμε σε μια ε, ζώνη που ήταν στο επίκεντρο της αναπλής σύγκρισης και πήγαμε και στο παρατηρητήριο ε, στα εργαστήρια ειρήνης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κολομβία, που λειτουργούν το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι. Και μάλιστα στην Bayern Pass βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια ειρήνη σε μια ζώνη ένοπλη σύγκρουση με τις ΦΑΡΚ. Και παρόλα αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά. Ένα από τα προβλήματα που ίσως επιδεινωθούν ε, στο μέλλον στην Κολομβία είναι η ασφάλεια. Γιατί από τη μια έχουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, από την άλλη όμως αυξάνονται ε, οι συμμορίες, οι εγκληματικές συμμορίες και αυτές οι συμμορίες, όπως είπε και ο κύριος Φίσας, αφενός προστατεύουν ε, την παράνομη εξόριξη ε, και ταυτόχρονα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Δημιουργούνται λοιπόν, ε, πολλαπλασιάζονται αυτές οι εγκληματικέ συμμορίες και δημιουργούν μια κατάσταση αστάθειας και έλλειψη ασφάλειας σε πολλές ζώνες της Κολομβίας εκεί που στο παρελθόν είχαμε παραστρατευτικέ και αντάρτικες οργανώσει. τώρα έχουμε και αυτέ τι εγκληματικέ συμμορίε που προστατεύουν τι παράνομε εξορίξει και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αυτό θα είναι σοβαρό πρόβλημα στην Κολομβία για το μέλλον. Οπότε όλε οι προσπάθειε των ελληνευτικών διαπραγματεύσεων επισκιάζεται από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ασφάλεια που ίσω δημιουργήσει ε, ακόμη μεγαλύτερε. Ε, ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον στην Κολομβία. Επίσης το θέμα των ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεων ε, που έχουν αρμοδιότητες από τους Δήμους και που ενημερώνουν τους Δήμους για τους εκτοπισμένους, για τους ανθρώπους που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Είναι άνθρωποι που θα πρέπει να εξάρουμε το έργο τους γιατί δίνουν καθημερινά μάχη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο Σανταντέρτο Κιλατσάου συναντηθήκαμε με έναν δήμαρχο ε, που μας ενημέρωσε για τις σχεδόν καθημερινές ανθρωποκτονίες που διαπράττονται και μάλιστα είχαμε επαφή και με ανθρώπους στα θύματα βίας και αυτοί οι άνθρωποι μας ε, θερμοπαρακάλεσαν να τους βοηθήσουμε για να συνεχίσουν τον αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί πραγματικά είναι οι αφανείς ήρωες της ε, Κολομβίας. Και όταν μιλήσαμε για τους υπερασπιστές και τους συνηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μερικές φορές τα λέμε συνηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκεφτόμαστε τις σημαντικές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά εκεί έχουμε και πραγματικά ε, τοπικές οργανώσεις που είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί ε, στέλνουν τους ανθρώπους τους ε, σε όλες τις ε, εμπόλεμες ζώνες της Κολομβίας και είναι οι αφανείς ήρωες που καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να, εξάρουμε το έργο τους σε αυτό το διαρθρωμένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε την Κολομβία. Θα πρέπει να τονίσουμε φυσικά την πρόοδο αλλά και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάστρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης που είναι η εκπόνηση του προπολογισμού της Ένωσης για το 2014. Ε, και πάλι ο κύριος Λάστρα είναι ο εισηγητής. Ε, σήμερα είστε πρωταγωνιστής κύριε Λάστρα. Σας δίνω το λόγο. Ναι, βλέπω ότι σήμερα εγώ έχω πολλή δουλειά, αλλά βλέπω ότι το ακροατήριο είναι ελάχιστο αλλά και τα θέματα των ε, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας ε, είναι πολύ σημαντικό και το γνωρίζει και ο κύριος Γκέρνς. Λοιπόν, ως προς τον προϋπολογισμό. Πριν από μία εβδομάδα λάβαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 και έχω πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τις αναφέρω στη συνέχεια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται από μια αναδιοργάνωση των δημοσιονομικών γραμμών και από πολλές αλλαγές που κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτες. Το επισημαίνω αυτό γιατί τα σχόλια δεν διευκολύνουν τις συγκρίσεις με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, κάτι που επιτείνει την έλλειψη διαφάνειας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό το 2014 ε, χαρακτηρίζονται από συγχώνευση γραμμών, από περικοπή κονδυλίων, αλλά κυρίως από ε, ε, προϋπολογισμούς που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και απορίες, που ελπίζω να μας τις επιλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα συνολικά ποσά, δυστυχώς το πιο κραβαλαίο στοιχείο της πρότασης είναι οι περικοπές των προϋπολογισμών που είναι σχεδόν οριζόντιες. Αυτό φυσικά αντιβαίνει τις ανάγκες που έχουμε σε ό,τι αφορά τις αναλυμένες μας υποχρεώσεις και τις ε, δραματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, για το μέσο ε, αναπτυξιακής συνεργασίας έχουμε μείωση 12,6% και για τις πληρωμές 10,7% λιγότερα κονδύλια από τη φέτος. Για την ανθρωπιστική βοήθεια έχουμε κάπως καλύτερη κατάσταση, 4,6% επιπλέον στις αναλήψεις υποχρεών, αλλά 4,4% λιγότερο στις ε, πιστώσεις πληρωμών. Οπότε διαρωτόμαστε γιατί τόσο δρακόντιες περικοπές και πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις ε, με τόσο πενιχρά κονδύλια. Κάτι που διαπιστώνουμε με ικανοποίηση είναι ότι αυξάνεται η ενίσχυση εκτάκτου ανάγκης. Προτείνεται ε, από 264 σε 296 εκατομμύρια ευρώ στις αναλήψεις υποχρεώσεων και από 80 σε 150 εκατομμύρια στις πιστώσεις πληρωμών. Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση του προϋπολογισμού και τα οριζόντια ζητήματα, η συγχώνευση κάποιων δημοσιονομικών γραμμών και η δυσανάλογη γεωγραφική ταξινόμηση αλλά και η δυσανάλογη θεματική ταξινόμηση και ε, η συγχώνευση κάποιων δημοσιονομικών γραμμών και ε, η δημιουργία υποκατηγοριών δημιουργεί προβλήματα, όπως στην περίπτωση του κονδυλίου για τη φτώχεια, για τη διακυβέρνηση και το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Δεν είναι διαφανής ο προϋπολογισμός και είναι δύσκολο και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες αλλά και να εξακριβώσουμε το κατά πόσο υλοποιούνται. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής που θα καταθέσουν τροπολογίες να διαβάσουν και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πολλά σημαντικά θέματα φαίνεται ότι παραλείπονται. Το 20% το, της βοήθειας θα πρέπει να πάει, από την, να θα πάει στην εκπαίδευση ή να υπόψη και οι ανάγκες της επικοινωνίας. Φαίνεται ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιμέρους αναλύσεις. Θα έλεγα ότι ότι είχαμε σημαντική μείωση του προπολογισμού για τη Λατινική Αμερική. Αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη μια σωστή λύση και δικαιολογία για το ποιες δραστηριότητε θα μειωθούν και τι θα γίνει προκειμένου να μην διακυβευθούν οι μέχρι τώρα προσπάθειες. Επίσης, ε, πώς οι κυβερνήσει θα αναλάβουν περισσότερες ευθύνε και πιστεύετε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τι παρατηρήσεις, γιατί δεν αναφέρεται η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, η υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ΜΚΟ, ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του εμπορίου και ε, των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δεν αναφέρεται ότι το 20% της βοήθειας θα πρέπει να δοθεί στις, στην παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών. Για την Ασία προτείνεται σημαντική αύξηση σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013. Αλλά δεν αναφέρεται ειδικό κονδύλιο για το Αφγανιστάν. Φαντάζομαι ένα τμήμα θα πάει στο Αφγανιστάν. Επίσης δεν υπάρχει καμία ένδειξη για τα σχέδια ως προς τη Βυρμανία Μιανμάρ και επίσης για τη γεωγραφική κατανομή των πόρων που προβλέπονται για την Ασία δεν, προβλε... δεν αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνολική ενίσχυση για την Ασία θα πρέπει να αυξηθεί ενώ η αντίστοιχη ενίσχυση για τη Λατινική Αμερική θα πρέπει να μειωθεί. Επίσης, ε, για να αυξηθεί το κονδύλιο για την Ασία, μειώθηκαν τα κονδύλια για άλλες περιοχές. Προς τι όλα αυτά. Στις παρατηρήσεις δεν αναφέρεται η σωστή κατανομή του εισοδήματος. Η σωστή ανακατανομή του εισοδήματος. Εύλογη απορία. Γιατί διαγράφηκε ο στόχος της βοήθειας των λιγότερο ε, εκπροσωπημένων ομάδων για να δοθεί μια φωνή και σε αυτούς αναφέρεται στο σχέδιο προϋπολογισμού η ανάγκη ε, να λάβουμε υπόψη τη μείωση της ενίσχυσης. Εδώ και πολλά χρόνια σημαντικά προγράμματα θα αφιερωθούν στη, στα προγράμματα διαχείρισης και καταπολέμησης των ναρκωτικών. Αλλά τα αποτελέσματά τους είναι αμφίβολα. Ε, το καθεστώς του Ουσμπεκιστάν είναι ιδιαίτερα καταπιστικό. Υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση και χυλάει η κυβέρνηση ε, κονδύλια παρά τις ε, συστηματικές επικρίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης έχουμε 33% της μείωσης των υποχρεώσεων. Πώς πιστεύετε ότι παρά τη μείωση αυτή θα υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά δυσίωνες. Γιατί ενώ έχουμε αναφορές για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, ε, της αξιοπρεπής απασχόλησης, της ισότητας ε, των ευκαιριών. Ε, για τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά για την Ασία δεν αναφέρονται οι στόχοι αυτοί, ενώ η στήριξη των ε, επιχειρήσεων ενέργειας προκειμένου να βελτιωθούν οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ασία είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται στην σχετική γραμμή. Βελτίωση της ασφάλειας και βελτίωση των διεθνών μεταφορών του ανεφοδιασμού σε ενέργεια και ή διασυνδέσεων των δικτύων και των φορέων τους. Επίσης, η νομοθετική, η κανονιστική και διοικητική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός στόχος, αλλά δεδομένου του πενιχρού υπολογισμού της ε, ε, αναπτυξιακής βοήθειας διακυβεύεται η υλοποίηση αυτών των στόχων. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, δηλαδή Ιράκ, Ιράν και η Ούτε ε, και εδώ υπάρχει σαφήνεια στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κονδύλια προβλέπει για τη Μέση Ανατολή και για ποιε χώρε. Και για την Νότια Αφρική έχουμε μείωση του ποσού. Και μάλιστα περιορίζεται η παροχή ενίσχυση στο θέμα της παιδείας. Και πάλι μας λείπουν πληροφορίες, τις οποίες ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια δημοσιονομική γραμμή με τα δημόσια αγαθά. Εκεί αναφέρει την επιστηστική ασφάλεια, το περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία, την ισότητα των φύλων, τα, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχουμε ένα γενικό κονδύλιο που είναι σαν μαύρο κουτί με 640 εκατομμύρια αλλά με μεγάλη διαφάνεια. Γι' αυτό και αποκαλώ αυτό το κονδύλιο ως μαύρο κουτί. Θέλω και εδώ διευκρίνηση. Πάλι, συγχώνευση των δημοσιονομικών γραμμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνδυάσει ε, τα κονδύλια για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και τους ε, μη κρατικούς φορείς. Εδώ αναφέρεστε στις τοπικές οργανώσεις κατά λάθο πιστεύω. Εξαιτίας της εσκεμμένης απαξίωσης του έργου των μη κρατικών δομών. Επίσης έχουμε 5-6% μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό. Τα κονδύλια ανθρωπιστικής βοηθείας μαζί με το θεματικό, αποθεματικό της εκτάκτου ανάγκης έχουμε μια ε, ε, ελάχιστη αύξηση παρόλο που και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχώνευσε τις γραμμές για την ανθρωπιστική επισητιστική βοήθεια και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των θεομηνιών. Ως εισηγητής θεωρώ ότι οι στόχοι μας ε, θα πρέπει να είναι εξή ε, και αυτό να προσέξουμε στις τροπολογίες μας. Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και να ε, μεγιστοποιήσουμε τα κονδύλια για την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια να δρομολογηθούν τα ποσά αυτά σε ζώνες όπου θα γίνει καλύτερη χρήση τους, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για άλλους στόχους. Σε ό,τι αφορά το μέτρο αναπτυξιακής συνεργασίας, θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των κονδυλίων στις διάφορες δημοσιονομικές γραμμές, χρησιμοποιώντας το περιθώριο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι 159 εκατομμύρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Με το ποσό αυτό δεν μπορούμε παρά να κάνουμε μικρές προσθήκες στις δημοσιονομικές γραμμές του μέσου ε, δημοσιονομικού ε, αναπτυξιακή συνεργασία που είναι 2 δι 250 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, οι προτάσει μα θα πρέπει να είναι συνεπεί με του στόχου μα ε, για τις διαπραγματεύσεις του κανονισμού DCI. Και εκεί θέλουμε το 60% της χρηματοδότησης να δίνεται στα γεωγραφικά προγράμματα, το 25% στα θεματικά προγράμματα, το 10% στις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές και το 5% σε ένα παναφρικανικό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το θεματικό σκέλος, υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες που μοιάζουν αλλά δεν συμπίπτουν με τις κατηγορίες των δημοσιονομικών γραμμών. Πιστεύω ότι είναι εύλογη η επιδίωξη ανάκτησης προηγούμενης ισορροπία μεταξύ Ασία και λοιπόν περιοχών του κόσμου και ιδιαίτερα με τη Λατινική Αμερική. Είναι επίση σαφέ ότι χάρη διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου θα πρέπει να αποκαταστήσουμε ε, κάποιες δημοσιονομικές γραμμές και η γραμμή για τα δημόσια αγαθά θα πρέπει να υποδιαιρεθεί αντικατοπτρίζοντας τις κατηγορίες του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας και θέλουμε ξεχωριστές γραμμές για τις μη κρατικούς φορείς και τις τοπικές αρχές. Αντίθετα, η συγχώνευση της ανθρωπιστικής με την επιστημιστική βοήθεια θα μπορούσε να γίνει δεκτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διορθώσουμε και κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια που γίνονται αποσαφηνίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι έγκυρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το 20% ε, ε, των στοιχειδιών υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλιστεί και να μην ξεχνάμε και τους στόχους που θέσαμε για το DCI ώστε να μην χαθούν αυτοί οι στόχοι. Τέλος, για τη διαδικασία. Είναι πραγματικά κρίμα που το τόσο σημαντικό αυτό έργο θα γίνει με τόσο ταχύς ρυθμούς και τόσο βεβιασμένα και στα πλαίσια της καθυστερημένη υποβολής τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2004 και της παράπολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο, φτάσαμε σε αυτή την πίεση του χρόνου και στην υποβολή ε, του Τη έκθεσή μας για τις 28 Αυγούστου. Α με διορθώσει η γραμματεία αν κάνω λάθος. Στο μεταξύ θα πρέπει να γίνουν οι μεταφράσεις και γι' αυτό ε, οι τροπολογίε μας θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι μέσα Ιουλίου. Έχουμε δηλαδή μόνο μία εβδομάδα για να συντάξουμε τις τροπολογίε μας. Και άρα η προθεσμία για τις τροπολογίες λύγει την επόμενη Τρίτη. Βέβαια, όπω πάντα, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να συντάξουμε την γνωμοδότησή μας. Αυτή δεν είναι τόσο ε, πιεστική. Θα προσπαθήσουμε πάντως για τη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου να έχουμε ετοιμάσει για να, και να έχουμε υποβάλει την γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα στους ευρωβουλευτές που το ζήτησαν. Ο κύριος Γκέρενς πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι ο συνάδελφος εισηγητή εστερνίζεται ένα μάθημα που έμαθα εγώ πριν από δύο χρόνια, όταν εγώ ήμουν εισηγητή. Ε, επέκρινα την Επιτροπή για έλλειψη φιλοδοξία και ε, ορκίστηκα να μην ξαναπέσω αυτό το λάθος και χαίρομαι που εστερνίστηκε το μάθημα και ο συνάδελφο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Με βάση τα στοιχεία που μας έχουν υποβληθεί, δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται η αρχή της διαφοροποίησης. Χρειάζεται λοιπόν μία προσέγγιση χώρα προς χώρα για να δούμε ποιες χώρες θα διαγραφούν από τον κατάλογο των ε, δικαιούχων. Δεύτερο σημείο, ο προϋπολογισμός αυτός εντάσσεται στα πλαίσια των συζητήσεων και της απόφασης που δεν έχει ακούσει ακόμα ληφθεί και αφορά το Multi-Financial Framework. Αναφέρεται ότι μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη Μεσολάβηση Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η ελαστικότητα θα πρέπει να γίνει κατανοητή σαν ένα αντιστάθμισμα για τα λιγότερα ποσά, για τα λιγότερα κονδύλια του Ταμείου. Θα ήθελα λοιπόν να με διαφωτίσετε για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε να γίνει μία προσωμείωση για να δούμε αν η ελαστικότητα στην περίπτωση που γίνει δεκτή θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πιστώσεων των χωρών μελών. Αυτό, των πιστώσεων πληρωμών και όχι δεσμεύσεων γιατί αυτό είναι μια διακόσμηση. Όταν εξαφανιστεί το χρώμα, η διακόσμηση παραμένει η ουσία που είναι πιστώσει πληρωμών. Θα μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο για να διαπιστώσει εάν οι διαπραγματεύσει που ε, έγιναν μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργούν ένα επιπρόσθετο ποσό. Γιατί πιστεύω ότι δεν ε, θα μπορούσαμε εξάλλου το ανέφερα αυτό Α, γίνεται πολύ συχνά αναφορά στη μόχλευση το θέμα είναι τι θα δοθεί στην ε, βοήθεια στην ενίσχυση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και πιστεύω ότι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί από το Συμβούλιο, ε, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Γιατί εάν η προσωμείωση στην οποία αναφέρθηκα θα μας μάθει ότι είναι αρνητική, δεν θα μπορούσαμε, δεν θα παραμείνει το πράγμα το έχουν ως προς την απόφαση που πρέπει να υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο. το Κοινοβούλιο έχει όλα τα ατού με, την, το μέρος του. Καταλαβαίνετε ότι θα πέσουμε και πάλι στον προπολογισμό του 2013 που μετά από την παρουσίαση από πλευράς του εισηγητή πιστώσαμε ότι είναι σαφώς υψηλότερος από αυτό που μας προτείνεται για το 2014. Εγώ πραγματικά δεν έχω τι να πω σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Ωραία. Ας δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κάρλο Άιτσα από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟΤ, κεφαλής ε, προγραμματισμού και προπολογισμού. Μπροστά σε αυτή τη χιονοστιβάδα ε, θεμάτων που ετέθησαν από τον κύριο εισηγητή και από τον κύριο Γκέρεντσα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι στα πλαίσια της νομοτολογίας του προπολογισμού που έχει δημιουργηθεί, κάναμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αν σας δίνουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, τότε έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαταστήσαμε τις δραστηριότητες statements όπως τις γνωρίζαμε με προγράμματα statements για να είναι πιο αντικειμενικός ο προπολογισμό και για να υπάρχουν δείκτες που θα μπορούσαμε να τους ακολουθήσουμε. Στο DCI και στο ENI θα πρέπει να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Θα πρέπει να συνδυάσουμε από τη μία πλευρά τη γεωγραφική πτυχή και από την άλλη πλευρά την θεματολογική και αντικειμενική πτυχή, ή σκέλος η απλούστευση, η απλοποίηση και αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι ότι καταρχάς όλες οι γραμμές που αφορούν τη συνεργασία βρίσκονται στον τίτλο 21 Ανάπτυξη και Συνεργασία και ε, μεταξύ του 19 και 21. Το δεύτερο είναι ότι όλες οι γραμμές που αφορούν ένα και μόνο μέσο βρίσκονται σε ένα κεφάλαιο και αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη ελαστικότητα και στην ε, περίπτωση ε, ανάγκης για κάποια διευθέτηση <clears throat> θα μπορούσαν πιο εύκολα να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά το TCI, η νομική βάση είναι η διαφορά μεταξύ του θεματικού και του γεωγραφικού προγράμματος. Ο βασικός στόχος είναι η μείωση της ένδυας και η οικονομική και κοινωνική και περιοριστική ανάπτυξη πρέπει να γίνει βιώσιμη και θα πρέπει να προωθηθεί η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλή διακυβέρνηση. Ε, Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή για την υποστήριξη της Παναφρικανικής Στρατηγικής δύο θεματικές γραμμές, Global Public Goods, Challenges, Civil Society, Local Authorities. Αυτές οι γραμμές υποδιαιρούνται στους δύο συγκεκριμένους υποστόχους. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά τις θεματικές γραμμές. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε περισσότερο με μεγάλα έργα που καλύπτουν <clears throat> τις διάφορες ε, πτυχές. Προσπαθήσαμε να κάνουμε και προγράμματα που παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα και στους διάφορους τομείς. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο προσπαθήσαμε να κινηθούμε. να κινηθούμε. Όπως διαπιστώνουμε, ο προϋπολογισμός του 2014 είναι πιο συρρυκνωμένος σε σχέση με του 2013. Απλά και μόνο γιατί είμαστε κινούμεθα στα πλαίσια του MFF. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε μια πρόταση παραμονών εκτός του MFF. Άκουσα την πρόταση του κυρίου Γκέρενς που είπε να επανέλθουμε στον προϋπολογισμό του 2013 Κοιτάξτε, δεν θέλω να εκφέρω άποψη. Αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Το δεύτερο που κάναμε, εφαρμόσαμε τη διαφοροποίηση. Δηλαδή να έχετε ένα κατάλογο των διαφόρων χωρών. Εμείς εφαρμόσαμε ένα μοντέλο για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις ανάγκες των διαφόρων χωρών στα πλαίσια της Agenda for Change και προσπαθήσαμε να δούμε αυτό το προϋπολογισμό. Αυτό οδηγεί σε μια ουσιαστική μείωση για την Λατινική Αμερική ιδιαίτερα σε επίπεδο διμερών προγραμμάτων που αντισταθμίζονται εν μέρη από μία αύξηση των περιφερειακών προγραμμάτων. Αυτό οδηγεί σε μία αύξηση υπέρ της Ασίας. Βεβαίως θέσατε μία σειρά από ερωτήματα ως προς το Αφγανιστάν που συμπεριλαμβάνεται στις γραμμές του προϋπολογισμού. Είναι μία συγκεκριμένη, συγκεκριμένο κονδύλι το οποίο αφορά το γενικό πλαίσιο της Ασίας. Βεβαίως υπάρχει και το Μπαγκλαντές που είναι μια φτωχή χώρα και θα πρέπει να υπάρξει μια μαζική κινητοποίηση. Αυτό αφορά συνεπώς τις δύο ε, δεσμεύσεις. Α, και, έχουμε και το μια μαρα. Αυτό αφορά την Κίνα, την Ινδία και αυτές τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Ασία, πιστεύω ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση σε σχέση με το φετινό προπολογισμό. Θέσατε και το θέμα που αφορά τους μη κρατικούς φορείς. Θελήσατε να κάνετε μια σαφή διάκριση όπως αυτή που αφορά δύο ξεχωριστά κονδύλια. Γιατί αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια πιο σφαιρική αντίληψη και να υπάρχουν προγράμματα που αφορούν διάφορα θέματα, όχι μόνο το περιβάλλον και το κλίμα, αλλά προγράμματα που έχουν στόχους που αφορούν τα διάφορα θέματα. Α, μισό λεπτό έχω κρατήσει μερικές σημειώσεις. Σε ό,τι αφορά την Αφρική πιστεύω ότι αναφέρεστε στη Νότιο Αφρική. Όντως υπάρχει μια σημαντική μείωση σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής ε, της διαφοροποίησης. Η Νότιος Αφρική είναι μια αναδυόμενη χώρα. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλα σας τα ερωτήματα. Ξέρω ότι καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να δώσετε απάντηση στα ερωτήματά μας, σχετικά και άσχετα ερωτήματα. Γιατί τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν και σχετικά και άσχετα. Εγώ θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς το... Για... Αν με ρωτήσει κάποιος για το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι να πω. Η Κολομβία θα διαγραφεί από τον κατάλογο των δικαιούχων. Και πάλι δεν έχουμε μια απάντηση. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα για το Παναφρικανικό ε, πρόγραμμα. Αν κάποιος μου θέσει το ερώτημα πώς ε, θα εφαρμοστεί η ελαστικότητα, δεν έχω απάντηση να δώσω. Πραγματικά νιώθω ηλίθιος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα. Ετέθησαν συγκεκριμένα ερωτήματα. Είστε έτοιμοι να προσωμιώσετε την ε, προσπάθεια αυτή ευελιξίας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν καταφέρουμε να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, Καταλαβαίνετε ότι θίγεται η ουσία αυτής της συμφωνίας της που θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Εγώ δεν έχω απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Απλά και μόνο θέτω ορισμένα ερωτήματα σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα δύσκολο. Να ξέρετε ότι πραγματικά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πάνε να προχωρήσουν τα πράγματα, να προχωρήσει ο προγραμματισμός. Παρόλες τις συζητήσει που είχαμε για τις ε, καταξουσιοδότηση πράξεις, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μην υπάρξει καμία κατάχρηση από πλευρά τη Επιτροπή και για να μπορέσει να δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκέρενς. Ξέρω, πιστώνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και για μας, γιατί και εμείς είμαστε υπόλογοι. Και στην Επιτροπή Ανάπτυξης όλες οι πολιτικές ομάδες έχουμε τις ίδιες προσδοκίες. Γι' αυτό και επιμένουμε σε αυτά που ζήτησε ο κύριος Γκόρενς, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για μας. Και μάλιστα τα θέλουμε το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι δυνατό να συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Ο κύριος Λάστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πράγματα είναι απλούστατα. Έχω απλώς να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στις ερωτήσεις μου. Αν θέλετε να τις στείλω και ηλεκτρονικά για να απαντήσει ελπίζω πριν την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προλάβω να συντάξω τις τροπολογίες μέχρι την επόμενη Παρασκευή και να είναι και λογικές οι τροπολογίες. Επιμένω, η συνένεση για την ανάπτυξη είναι το βασικό θέμα και όχι η το θεματολόγιο για την αλλαγή. Η συνένεση για την ανάπτυξη. Και αν το ε, επιχείρημά για την αύξηση του κονδύλου της Ασίας είναι η Κίνα γιατί δεν χρησιμοποίησατε αντίστοιχο ε, επιχείρημα και για τη Λατινική Αμερική που και εκεί η Κίνα έχει αυξήσει την παρουσία της. Επαναλαμβάνω, δεν έλαβα καμία απάντηση, θα στείλω τις ερωτήσεις μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις ε, περιμένω απαντήσεις το συντομότερο δυνατό για να προλάβω να συντάξω και τις τροπολογίες μου. Καλώς. Περιμένουμε απαντήσει το συντομότερο δυνατό. Τροπολογία για την κατάθεση των απολογιών. 17 Ιουλίου, Τετάρτη, το μεσημέρι. Όπως είπε και ο συγητής, θα ετοιμάσουμε και γνωμοδότηση ε, που θα δώσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα εξετάσουμε τη γνωμοδότησή μας στη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση ραντεβού στις 3 το απόγευμα, 3 σε παραλαμβάνω και όχι 3 και 4 όπως είχε αναγγελθεί αρχικά. Γιατί προσθέσαμε και μία σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον αντιπρόεδρο του Μπουρούντι μετά από αίτημα του συναδέλφου Λουί Μισελ. Καλή σας όρεξη λοιπόν και ε, σας περιμένω με το απόγευμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.